Mesdames et messieurs, θα συνεχίσουμε Θα ήθελα να κάνω την εξή διευκρίνηση. Μετά από την απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής μας, προβλέψαμε ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες της έκθεσης Βένσον για το εμπόριο και την ανάπτυξη που θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα, ανταλλαγή απόψεων που θα κάνουμε σήμερα το πρωί μετά το σημείο 13. Πρόκειται για παρουσίαση μελέτης για τα ε, τη της βιοτεχνολογίας αναπτυσσόμενες χώρες. Θα εξετάσουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Αργεντίνη για ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, Κεντρικής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της ουσίας είναι η συντάκτρια γραμμοδότησης, κυρία Σαρτζεντίνη, θα πάρει αμέσω το λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σύντομη η γνωμοδότησή μου. Μία φράση στην οποία λέγεται η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αρμόδια επί της ουσίας να αρνηθεί να εγκρίνει τις συμφωνίες αυτής ε, της ενδιάμεσης με το Καμερούν. Το να μπει, μπει κανείς όχι σε κάτι το οποίο νομίζουν ε, όλοι πρέπει να πει είναι ίσως οδηγήσει σε παρανόηση, αλλά πρέπει να πω ότι πριν από δύο εβδομάδες είχαμε και εγώ ήμουν επίσης εισηγήτρια το παρεμφερές με για την Νότια Αφρική και συμφωνήσαμε με την απόψή μου όλοι οι συνάδελφοι ότι δεν θα πρέπει να επικαιρώσουμε αυτή την ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Σήμερα για άλλους λόγους λέγω να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική. Μιλούμε για ένα κράτος της Κεντρικής Αφρικής, το Καμερούν, και νομίζω ότι υπάρχει μόνο μία περιφερειακή τέτοιου συμφωνία το Καμερούν έχει γειτονικέ χώρε οι οποίε κάποιε από αυτέ τι έχουν διαφορετική άποψη. Άρχισαν οι διαπραγματεύσει το 2007 και η Εθνοσυνέλευση του Καμερούν ακόμη δεν έχει επικυρώσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω εμείς να περιμένουμε. Υπάρχουν κάποια μήνυματα από το Καμερούν ότι θέλουν να αναθεωρήσουν κάποια μέρη της ενδιάμεσης αυτής συμφωνίας, κυρίως αυτά που αφορούν την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά του Καμερούν και την απελευθέρωση το 80% των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιμένουμε λίγο. Στην γνωμοδότησή μας προς την ΙΤΑ δεν υπάρχει αυτή η παρατηρήση. Γι' αυτό ζητώ να καθυστερήσουμε την επικύρωση, ώστε να δώσουμε στο Καμερούν την δυνατότητα να αναθεωρήσει το όλο θέμα. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε, δεδομένου ότι και από την άλλες πλευρά δεν έχει υπάρξει επικύρωση. Θα δούμε όλο και περισσότερες ενδιάμεσες συμφωνίες οικονομικές εταιρικέ σχέσεις στο εγγύς μέλλον και το πρόβλημα είναι ότι ενώ αυτό είχε θεωρηθεί ως ένα μέσον ανάπτυξης, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και δεν βοηθούμε την κατάσταση για την ανάπτυξη και υπονομεύουμε ακόμη και το ε, όλο θέμα της ε, αναπτυξής της περιοχής. Εάν αρχίσουμε να συνάπτουμε και να επικυρώνουμε τέτοιους ε, ενδιάμεσες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής ε, σχέσεις με κάποιες χώρες. Ο ΤΕΙΣ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι ο Νόρμπερτ Νόης μαζί μας ακόμη γιατί λόγω μιας απεργίας στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης ε, έμεινε εκεί και έτσι θα διαβάσω εγώ το κείμενό του. Λοιπόν, τα έξι σημεία έχει σημειώσει και θα σας τα διαβάσω εγώ. Λέει Νόμπερτ, ευχαριστώ την κυρία Σαργεντίνη για το σχέδιο έκθεσή τη. Κάποιε από τι ανησυχίε τη καταλαβαίνω σχετικά με την προσωρινή συμφωνία, αλλά δεν συμφωνώ με το συμπέρασμά τη. Όπω όλοι γνωρίζουμε, η τωρινή κατάσταση δεν είναι συμβατή με τον ΠΟΕ και η πρόσβαση στην αγορά που έχουμε τώρα δεν θα διαρκέσει για πάντα. Αναγνωρίζω το πρόβλημα ότι πολλέ χώρε στην περιοχή τη Κεντρική Αφρική είναι από τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και επωφελούνται από την πρωτοβουλία, από του κανόνε όλα από Αυτές οι χώρε λοιπόν δεν έχουν κίνητρα να διαπραγματευτούν μια τέτοια συμφωνία εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδιε χώρε όμω δεν θα μείνουν λιγότερο ανεπτυγμένες χώρε για πάντα και τελικά θα υπογράψουν και αυτέ μια τέτοια συμφωνία αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να μας εμποδίσει να ασχοληθούμε με τη συμφωνία αυτή που έχει διαπραγματευτεί και υπογράψει το Καμερούν παρότι δεν την έχει επικυρώσει ακόμη διότι το Καμερούν δεν είναι μία από τις χώρες ε, του καθεστώτος όλα εκτός από όπλα και χρειάζεται μία εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο σημείο πρέπει να υπάρξουν αντισταθμίσεις ε, τουλάχιστον ε, κατά το χρόνο που απαιτείται για την μεταρρύθμιση του εσωτερικού συστήματος φορολογίας του Καμερούν. Το Καμερούν θα υποφεληθεί από ένα σύστημα, καλύτερο φορολογικό σύστημα μακροπρόθεσμα ούτως ή άλλως. Αυτά είναι τα σημεία του Νόμπελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μίτσελ. Πρόεδρε, καταλαβαίνω αυτό το οποίο προτείνει η Judith, αλλά θα ήθελα να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Τι μας προτείνει να σταματήσουμε τώρα και να κάνουμε ε, την έγκριση στο μέλλον κάποια στιγμή. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό το σημείο λίγο καλύτερα. Τι ακριβώς μας προτείνετε. Δεν προτείνετε να τους βγάλουμε κόκκινη κάρτα, μάλλον κίτρινη κάρτα. Σωστά σας καταλαβαίνω. Κυρία Σαργεντίνη. Αυτές είναι οι καταληκτικές μου παρατηρήσεις. Ε, θα μου δώσετε το λόγο ξανά στο τέλος. Ναι, ναι, ναι, θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή και μετά θα κλείσετε με, τις, με την τελική σας παρέμβαση. Ναι, κύριε Μίτσελ, έχετε δίκιο. Με τη συζήτηση που κάναμε την τελευταία φορά, για την διάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, με χώρες της Αφρικής. Ε, προτάθηκαν κάποιες τροπολογίες από τους σοσιαλιστές ε, με σκοπό να παγώσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μια προφορική τροπολογία και δεν υπήρχε πλειοψηφία στην Επιτροπή και δεν πέρασε αυτή η τροπολογία και συνεχίσαμε με την δική μου πρόταση που ήταν να μην το επικυρώσουμε συνολικά. Παρ' όλα αυτά, έλαβα υπόψη μου την πρόταση των σοσιαλιστών που μας είπαν ας το παγώσουμε προς το παρόν, ας το αναβάλουμε και είμαι πρόθυμη να επανεξετάσω αυτή την πρόταση γιατί εξυπηρετεί το στόχο μου. Ο δικός μου στόχος είναι να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο Καμερούν, να δούμε αν θέλουν να την επικυρώσουν τη συμφωνία, γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μάλλον δεν θέλουν τώρα με τις τωρινές συνθήκες να κάνουν την επικύρωση. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έγγραφο αυτό. Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση με το Καμερούν είναι η αρχή μια ευρύτερη εταιρική σχέση με όλη την περιφέρεια. Επομένω, είναι μια προσωρινή λύση που θα επέτρεπε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσει για να έχουμε μια περιφερειακή συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση. Αυτός είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κεντρική Αφρική. Το Καμερούν όμως ε, τη χρειάζεται αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, γιατί χωρίς τη συμφωνία αυτή το Καμερούν θα έχει σοβαρές δυσκολίες για πολλά από τα εξαγωγικά του προϊόντα προς την Ευρώπη, που δεν καλύπτονται ούτε από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που είναι οι μπανάνες και το αλουμίνιο, τα προϊόντα αυτά τα εξαγωγικά μεταξύ Με τη συμφωνία αυτή από το 2008 το Καμερούν έχει διατηρήσει σημαντικούς τομείς της οικονομίας του και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Όσο για τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση, για τους οποίους προτείνεται να αρνηθούμε τη συμφωνία μας, η δική μας άποψη είναι ότι αυτή η ενδιάμεση συμφωνία δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε στην βιομηχανία του Καμερούν, ούτε στα κυβερνητικά έσοδα, ούτε στην περιφερειακή ολοκλήρωση. Και αν μου επιτρέπετε θα παραθέσω και κάποιους ε, λόγους για το επιχείρημά μου αυτό. Σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς το Καμερούν έχουν ε, αποκλειστεί, έχουν εξαιρεθεί ούτως ή άλλως γύρω στο 20%. Και ούτως ή άλλως η συμφωνία περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα 15 ετών, άρα επιτρέπει να παρέλθει ο χρόνος τον οποίο χρειαζόμαστε, χρειάζεται το Καμερούν για να κάνει τις προσαρμογές. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι ενδιάμεσα προϊόντα που χρειάζονται οι τοπικές βιομηχανίες στο Καμερούν. Είναι προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες του πληθυσμού του Καμερούν, όπως φάρμακα ή ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός. Και παράλληλα έχουμε και ρήτρες διασφάλισης στη συμφωνία που επιτρέπουν στους εταίρους μας να διακόψουν το προτιμησιακό καθεστώς που μας παρέχουν σε περίπτωση ανάγκης. Και αυτό περιλαμβάνει και τη ρήτρα για τις αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Υπάρχει επίσης ε, και το τμήμα της συμφωνίας που προβλέπει τεχνική και οικονομική βοήθεια, ιδίως για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Και συμφωνώ με το σχόλιο που έγινε ότι χώρες όπως το Καμερούν χρειάζονται φορολογική μεταρρύθμιση, γιατί θα πρέπει από το εμπόριο να περάσουν ε, στη φορολογία ως σύστημα ε, εσόδων. Όμως, ε, έχουμε σύστημα που μας βοηθά να βοηθήσουμε καλύτερα τη χώρα μέσω αυτών που προτείνουμε στη Συμφωνία. Και επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και ενδοπεριφερειακό εμπόριο, 2 με 3% και τα εμπόδια, όπως γνωρίζουμε, έχουν μεγαλύτερη σχέση με άλλα εμπόδια, όπως είναι η διαφθορά. Ζητήματα δηλαδή που θέλουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε. Μη δασμολογική φραγμή δηλαδή. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε πόρους στις περιφερειακές αυτές διαπραγματεύσεις για να περάσουμε σε μια πραγματικά περιφερειακή λύση, ενώ αυτό που έχουμε εδώ είναι μόνο η αρχή. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι οι διαπραγματεύσεις για την ενδιάμεση συμφωνία ολοκληρώθηκαν το 2007. Το Καμερούν τώρα προχωρεί προς την επικύρωση της συμφωνίας Η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά που τους δίνουμε είναι κάτι για το οποίο χρειάζονται την ενδιάμεση συμφωνία και ελπίζω να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέρμαν. Μια μικρή ερώτηση για την, για την Επιτροπή θα ήθελα να κάνω, αν το επιτρέπετε. Από τις 17 Δεκέμβρη του 2007, τότε που υπέγραψε η κυβέρνηση του Καμερούν. Είχατε, είχατε επαφές με την κυβέρνηση του Καμερούν και γιατί όχι. Αν ναι, τότε ποια είναι η εκτίμηση που, ε, που γίνεται όσον αφορά την επικύρωση από το Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας. Εκπλήσωμε, διότι περάσαν πέντε χρόνια από τότε θα, θα έπρεπε δηλαδή να καταλάβουμε γιατί ακόμα το Κοινοβούλιο δεν έχει βιαστεί να επικυρώσει. Πρόεδρος, μπορείτε να απαντήσετε σύντομα. Μιλάμε για το Κοινοβούλιο του Καμερούν. Υπάρχουν ίσως τρία σημαντικά πράγματα πριν να αναφέρουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, όλοι συνεχίζουν να στοχεύουν στην επίτευξη περιφερειακής λύσης, ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί αρκετά σύντομα μετά τη σύναψη αυτής της προσωρινής συμφωνίας, της ενδιάμεσης. Και με αυτό το πνεύμα αρχίσαμε να δίνουμε την ελεύθερη πρόσβαση στο Καμερούν ακόμη και πριν επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Πρώτη παρατήρηση. Τώρα, Δεδομένου ότι συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση, η ελεύθερη πρόεδρος του Καμερούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και με την ε, πρόοδο που υπήρξε σε περιφερειακό επίπεδο, είπαμε ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, το θέμα του κανισμού της πρόοδος στην αγορά, ελπίζουμε ότι θα επιληθεί σύντομα ώστε να υπάρχουν επιπτώσεις για το Καμερούν. Αλλά όσο η κατάσταση έχει ως εξής, δηλαδή ελεύθερη πρόσβαση και όχι ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, κανένας δεν βιάζεται να το ολοκληρώσετε. Και εμείς πέντε χρόνια μετά Περιμένουμε ακόμη την επικύρωση και ελπίζω ότι θα τους ε, ε, οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Σαργεντίνη για να ολοκληρώσουμε. Η άποψή μου στο ερώτημα που θέσατε κυρία Μπέρμαν είναι ότι επαφές μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Κατανοώ γιατί ε, στις χώρες αυτές ε, υπάρχουν ε, ε, οι διαπραγματεύσεις που ολοκληρώνονται μεταξύ Κομισιόν και ε, κυβερνήσεων. Δεν χρειάζεται πάντα επικύρωση, αν και από τα κοινοβούλια νομίζω ότι αυτό είναι ένα θεσμένο. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση για το Καμερούν. Διαβάσετε τα σχόλια και του συναδέλφου σας Νόισερ, που όντως ε, έκαναν ε, την διαπραγμάτευση για αυτή την ενδιάμεση συμφωνία. Αλλά, βεβαίως, όπως λέει και η Κομισιόν, χρειάζονται κάποια συμφωνία για να μπορούν να κινούνται στα πλαίσια των κανόνων του ΟΠΕ. Διαπραγμάτευση δεν σημαίνει ότι πάντα συμφωνείτε με το αποτέλεσμα. Και εάν δούμε πώς έχουν τα πράγματα και εμείς τρενάραμε κάπως γιατί ελπίζαμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει τελικά αυτή η περιφερειακή συμφωνία και βεβαίως αυτό το τα πάντα εκτός από όπλα είναι Καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Χρονοτριβήσαμε λοιπόν. Εμείς όμως είμαστε από την πλευρά αυτών που επίσης διαπραγματεύσουν. Και αυτό το οποίο είναι προβληματικό είναι ότι προσπαθούμε όσο περισσότερο η Ήπειρος αυτή προσπαθεί να αναπτυχθεί να είμαστε εκεί και συγχρόνως να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη εμπορική συμφωνία με ελευθερικό στην αγορά. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι το 80% είναι χαμηλό ποσοστό. Είναι υψηλό θα έλεγα. Όταν μιλούμε για άλλε χώρες της ε, ε, νότιο-ανατολικής Αφρικής υπήρχαν ε, ποσοστά που δεν ξεπερνούσαν το 70, αλλά είναι καλό το 80. Και βεβαίως δεν είναι σωστό να λέγεται ότι εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε την ε, επικύρωση αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας με το Καμερούν. Επαναλαμβάνω, πρέπει να τηρήσουν και τους κανόνες του ΠΕ. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για το Καμερούν, το αναγνωρίζω, αλλά είναι εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τελικά να γίνεται καλύτερο μπορεί για το Καμερούν. Τελική παρατήρωση. Η πρώτη τέτοιου είδου ενδιάμενη συμφωνία έγινε με τις χώρες Καραβικής και μετά από δύο χρόνια έκαναν τις διαπραγματεύσεις και κατέληξαν ότι δεν πρόκειται για καλή συνοφία και στην τελευταία ε, κοινοβουλευτική συνέλευση το θέμα αυτό συζητήθηκε και Ευρωπαϊκή Ένωσης και μας είπαν ότι δεν τους ικανοποιούσε αυτή η ενδιάμεση συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα πρέπει η Κομισιό να παρατείνει τους κανόνες ε, πρόσβαση στην αγορά έτσι ως έχουν και να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία. Πολύ καλά. Πριν να ολοκληρώσουμε στο θέμα αυτό, επιτρέψτε μου να επενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάσταση τροπολεόνιων για την γνωμοδότηση είναι 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, ανταλλαγή απόψεων για την μελέτη που αφορά τον αντίκτυπο της βιοτεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, κυριότερη από τις οποίες είναι η ασφάλεια των, της διατροφικής αλυσίδας. Πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα δεδομένου ότι η δημογραφική εξέλιξη είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μέσα που διαθέτουν, περιορισμένα διότι υπάρχουν ε, προβλήματα με την επιδείνωση του περιβάλλοντος, δεν βοηθούν οι τεχνολογίες κτλ. Πολλοί πιστεύουν ότι οι γενετικά τροποποιημένες ε, τα γενετικά τροποποιημένα είδη διατροφής και καλλιέργειες είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει να λύσουν το πρόβλημα. Κάποιες χώρες, κάποιες άλλες πιστεύουν ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανικοί όχι δε μόνο δεν εγγυούνται τη βιοπικιλότητα, αλλά την επιδεινώνουν και την βλάπτουν. Αυτή η μελέτη λοιπόν καταρχάς θα παρουσιαζόταν από την τον κύριο Κάρσιν, ο οποίο για λόγους υγείας απουσιάζει, η κυρία Γκέστετερ από το ίδιο θα παρουσιάσει το θέμα. Όπως ελέγχθη, σας παρουσιάζω ε, σύντομα η μελέτη που σας ζητήσετε. Ασχολήθηκα όχι με το συγκεκριμένο θέμα εδώ, αλλά με παρεμφερεί θέματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω συνοπτικά να σας παρουσιάσω λοιπόν τα αποτελέσματα. Όπως ελέγχθη ήδη στην εισαγωγική παρατήρηση, η, τα γενικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι κάπως αμφιλεγόμενο θέμα. Θα πω λοιπόν τα εξή. Αν αρχίζει κανείς να δει τις μελέτες που υπάρχουν για το θέμα αυτό και τις επιπτώσεις οικονομικές και στην υγεία, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές αντιφατικές απόψεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε αξιόπιστα συμπεράσματα και έγκυρα κυρίως. Τρία θέματα άπτονται του θέματος αυτός και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν μιλούμε για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, τις μακροπρόθεσμες ε, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις που έχουν στην πραγματική ζωή, πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει αντικείμενο ε, εκτενών μελετών Μόνο εδώ και 15 χρόνια έχουμε τέτοιου είδους ε, τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά και είναι πολύ μικρός ο κύκλος αυτός. Δεύτερον, οι οικονομικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων τροφών είναι δύσκολο ε, να εξεταστούν διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές που υπησέρχονται και δεν μπορούμε να απομονώσουμε εύκολα από μεθοδολογικής πλευράς τις επιπτώσεις τους. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι ε, μεμονωμένα αν θέλετε, διαφορετικά για κάθε περίπτωση και υπάρχουν και διάφορα διαπλεκόμενα συμφέροντα μεταξύ εταιριών, αγοραστών, πολιτών Και πολλές φορές οι επιλογές οφείλονται σε άλλου είδους ε, ε, παρατηρήσεις. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις απλές και αξιόπιστες. Τώρα, πώς άρχισε η όλη συζήτηση και το όλο θέμα αυτό. Δεδομένου ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσμός, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φτώχειας, ε, ότι υπάρχουν ε, διατροφικές ε, κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ότι η κλιματική αλλαγή επίσης επηρεάζει την όλη κατάσταση και αν προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των γενικά τροποποιημένων στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να ωφελήσουν κυρίως τους ε, ε, φτωχότερους και τους μικρούς παραγωγούς και αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τι συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2011 160 εκατομμύρια εκτάρια είχαν καλλιεργηθεί με τέτοιου είδους ε, ε, προϊόντα σε 29 χώρες και ως σύγκριση θα σας πω ότι η καλλιεργούμενη επιφάνεια αν ε, σε ολόκληρη τη γη είναι της τάξης των 180 εκατομμυρίων. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προϊόντα τα οποία δυναμικά έχουν μπει σε όλες τις παγκόσμιες αγορές, η σόγια, το καλαμπόκι, το βαμβάκι και η... modified crops. Uh, one is um, the so-called BT um, crops that have an... κανόλα. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε herbicide tolerance, which means that you can treat them with herbicide and all the weeds will die, but the Και το κραμβέλαιο, το τέταρτο προϊόν, το οποίο έχει κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές. Θα πρέπει να αναφέρουμε ε, επίσης ε, το γεγονός ότι για τα προϊόντα αυτά ε, χρησιμοποιούνται οκτώνα. Υπάρχουν χώρες ε, αναπτυσσόμενες και φτωχές, οι οποίες έχουν κατακλειστεί από τέτοιου είδους γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Τώρα, ποιες είναι οι δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση τέτοιων προϊόντων. Ε, Το πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες είναι διαφορετικό από ό,τι για τις ανεπτυγμένες όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις υπάρχουν λοιπόν διαφορές, υπάρχουν ε, σε σχέση ε, με τα μη γενετικά τροποποιημένα προϊόντα διαφορές, υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση. Ε, μεγαλύτερη αντίσταση στα ζυζανιοκτώνα και στις διάφορες ασθένειες. Χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Ε, ανθίστανται καλύτερα στα διάφορα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Ε, λέγεται ότι χρειάζονται λιγότερα ε, εργατικό κόστος και ενεργειακό και κάποιοι πιστεύουν ότι όπως απέδειξαν και κάποιες μελέτες που δεν είναι πάντα όμως σαφείς που αφορούν την ε, εργασία, τα εργατικά χέρια που χρειάζεται. Άλλοι πιστεύουν ότι βεβαίως ε, έχουν ε, καλύτερη τιμή στην αγορά, αλλά βεβαίως ε, όλα εξαρτώνται από το προϊόν. Και βεβαίως άλλοι λέγουν ότι έχουν μεγαλύτερη διατροφική αξία. Τώρα, από την άλλη μεριά, είναι ακριβότερο οι σπόροι για τέτοιου προϊόντα. άρα υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από τους φορείς που τους διαθέτουν στο εμπόριο. Και είναι πιο απλό να έχει κανείς του δικού σπόρους παρά να προμηθευτεί τέτοιους. Επίσης, από ό,τι έχουν αποδείξει οι μελέτες, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη ποιες είναι μακροπρόθεσμα οικονομικές επιπτώσεις. Όπως σας είπα, στην αγορά κυρίως έχουμε τέτοιου είδους, ε, είδους ε, προϊόντα. Δεν ξέρουμε πώς ε, θα, θα είναι οι αλλαγές που θα υπάρχουν μακρονομικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, ίσως στο μέλλον θα υπάρξει ναι, ε, αλλαγή στον τόπο με τον οποίο αθίστανται τέτοιου είδους σπόροι και προϊόντα ε, στα διάφορα ε, προβλήματα και ζυζάνι θα χρειαστούν περισσότερα φυτοφάρμακα. Και όπως σας είπα δεν έχουμε γενικότερα αποτελέσματα. Τώρα, ποιοι τι επηρεάζει την ε, οικονομικές επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση των ε, γενετικά τροποποιημένων τροφίων. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά την ε, μέγεθος της εκμετάλλευσης, το κατά πόσον έχουμε να κάνουμε με ε, σπόρους οι οποίοι ανταποκρίνονται καλύτερα στο περιβάλλον της ε, εκμετάλλευσης. Η υποστήριξη που μπορεί να έχει και η επιδότηση ε, ένας ρώτες εξαρτάται από κατά πόσον είναι κάτι το οποίο γίνεται γενικά τρόπο στην Κίνα περιπίν, αυτά σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο πρέπει να δει κανείς κατά πόσον υπάρχει ε, διάθεση στην αγορά τέτοιου είδους προϊόντων, κατά πόσο σε διεθνές επίπεδο μπορεί κανείς να αναπτύξει συνεργασίες για την εξαγωγή τέτοιου είδους προϊόντων, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα και τα προϊόντα αυτά. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τους γεωργούς, αλλά ακόμη αγνοούμε πάρα πολλά θέματα που από τον αφού του γεγονότος και όπως είπα και προηγουμένως, εκεί που μέχρι τώρα καλλιεργηθεί τέτοιου είδους προϊόντα σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι και οι πιο φτωχές. Τώρα, να δούμε τι σημαίνει σε επίπεδο τιμών. Αυτό δεν ήταν μέσα στην αρχική παρουσίασή μου, αλλά μου ζητήθηκε να κάνω κάποια σχόλια και θα προτείνω αυτά τα οποία βρίσκονται σε στάδιο της μελέτης αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της προώθησης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τα θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ε, είναι ε, στοιχεία πρόσφατα και με πολλά κενά και όχι πάντοτε βάσιμα. Και σε αυτό το οποίο μου ζητήθηκε να πω, μια γενικότερη προοπτική έπρεπε να αναφέρω Το δεύτερο σημείο είναι οι επενδύσεις ε, στην έρευνα στο δημόσιο τομέα για να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιστηστικές ανάγκες στις αναπτυσσόμενες χώρες με βάση προϊόντα που καλλιεργούνται σε αυτή την, ε, τη χώρα. Τώρα, ε, τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ε, δεν είναι τα προϊόντα τα οποία ε, αποτελούν τα βασικά είδη διατροφής. Ε, είναι είδη όπως το κραμβέλαιο κανόλα που αναφέραμε προηγουμένως. Και το τρίτο σημείο είναι ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, διότι δεν γνωρίζουμε αρκετά θέματα αυτή τη στιγμή και γιατί υπάρχουν και πολλά αντιπαρατηθέμενα συμφέροντα σε αυτή τη συζήτηση. σε κάποιο βαθμό υπάρχει έλλειψη επιστημονικής γνώσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες, αλλά δεν υπάρχει επιστημονική συνένεση για το θέμα αυτό. Και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει την αρχή της προφύλαξης και αυτό νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί την χάραξη πολιτικής αυτή τη στιγμή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Τέλος, στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικό θέμα αυτό και η επίπτωση των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εξαρτάται και από τις τιμές των σπόρων και από το αν οι παραγωγοί μπορούν να ανταλλάσσουν σπόρους και να καλλιεργούν τους δικούς τους σπόρους και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να συνεισφέρει στην όξυνση αυτής της νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες με διμερείς εμπορικές συμφωνίες για να μην παρεμποδιστούν οι αγρότες να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία στο μέλλον. Αυτά προσπαθώντας να δώσω μια πολύ σύντομη παρουσίαση για αυτά που μου ζητήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω θα πιέζω λίγο, αλλά είμαστε καθυστερημένοι. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ όλοι να είναι κάπως σύντομοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη. Κωστέ, κύριος Κορτές Λάστρα θα πάρει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια της προφορία που μας έδωσε, που είναι Συμπληρωματικέ σε σχέση με την έκθεση της ΦΑΟ που έχουμε για την κατάσταση της γεωργία και την διατροφή το 2012. Στην ε, κύριος ε, Ναβάρο μας είπε ότι υπάρχουν και υπάρχει μια τρίτη επιλογή μεταξύ των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και την οικολογικών προϊόντων. Υπάρχει τρίτος δρόμος, όχι λιγότερο κυρίως, αλλά όπως είπε και η συγγήτρια, μελετώντας ε, την ε, κάθε καλλιέργεια, το κάθε έδαφες, ώστε να μπορέσουν να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την διατροφή όλο και περισσότερων ατόμων. Πιστεύω ότι το... και εσείς το την υπόψη. Το ερώτημα όμως σας είναι διαφορετικό. Τη Ρώμη στην Επιτροπή Επισητιστικής Ασφάλειας είδαμε και κάποιους εκπροσώπητες και τους κάναμε το εξή ερώτημα. Όταν πρέπει εσείς να δώσετε τρόφιμα, δίδετε γενετικά τροποποιημένα, μας είπαν ναι βεβαίως. Και μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στους λαούς στους οποίους δίδανται τέτοιους τρόπους. Βεβαίως πάντα υπάρχει το ερωτηματικό όσον αφορά τέτοιου είδους καλλιέργειες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Όσον αφορά την διατροφική αξία αυτών των τροφίμων, αυτών των προϊόντων, που διανέμονται στα πλαίσια της πληθυστικής βοήθειας ή μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Η κατανάλωση τέτοιου είδους ε, προϊόντων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, και το είδαμε αυτό για ένα-δύο χρόνια στην περίπτωση της ε, επιστημικής κρίσης που υπήρχε ο Σαχέλ ή αλλού. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα, το παγκόσμιο πρόγραμμα παροχής επιστημικής βοήθειας τέτοιου τρόφιμα προβλέπει, τι ε, απάντηση έχετε να μου δώσετε. Η Κομισιό θέλει να λάβει το λόγο, εάν όχι, η κυρία Γκέστέτερ για να απαντήσει. Θα, απαντήσω στην ερώτησή σας ε, για τις επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην υγεία. Δεν ήταν στο πλαίσιο της ενημέρωσης που θα έπρεπε να κάνω, αλλά μπορώ να σας δώσω μια γενική εικόνα των όσων γνωρίζω επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, εγκρίνει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για την κατανάλωση αυτό συμπεριλαμβάνει και μία αξιολόγηση επιπτώσεων ε, για την υγεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Τροφίμων για να ε, εγκριθούν αυτοί οι οργανισμοί που δεν έχουν επιπτώσεις επί της υγείας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για την επιστημιστική βοήθεια σημασία έχει το τι την κάνουμε. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά όταν δίνουμε επιστηστική βοήθεια για κατανάλωση ή σπόρους προσφορά, γιατί εκεί μπορεί να έχουμε και περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες και επιπτώσεις. Αυτό το οποίο θα με ενησυχούσε εμένα στην επιστηστική βοήθεια είναι ότι είναι θέμα επιλογής και τα τελευταία χρόνια κάποιοι από τους λαμβάνοντες επιστηστική βοήθεια μας έχουν πει δεν θέλουμε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Έχουμε κάποιες ανησυχίες, επομένως ε, πρέπει να δούμε κατά πόσο οι χώρες δωρητές το τηρούν αυτό. Αν είμαστε όμως σε μια κατάσταση όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη για φαγητό, μπορεί να δίνεται επιστημιστική βοήθεια για σύντομο χρονικό διάστημα Οπότε θα έλεγα ότι οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν ή που κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχουν ίσως δεν είναι τόσο σοβαρές γιατί δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων. Αλλά όπως σας είπα χρειάζονται μελέτες για να δοθεί μια προσεκτική απάντηση. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή για να μας δώσετε τόσο χρήσιμες πληροφορίες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Άρα προχωρούμε τώρα. Αμ, η ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση Σβένσον, το ξέχασα αυτό. Μήπως θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Σβένσον, παρακαλώ. Σβένσον. Σβένσον. Euh, σύντομα, αν γίνεται, κύριε Σβένσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξαφνικά έγινε αυτό. Και δεν υπάρχει στην μερίσια διάταξη αλλά μου προτάθηκε να πάρω αυτή την ευκαιρία για να εξηγήσω κάπως τις θέσεις μου για την, ε, τον κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν είναι πολλοί συνάδελφοι εδώ. Δεν είχε αναφερθεί το θέμα μου στη μέση διάσταξη δυστυχώς. Όσον αφορά τις ε, παραγράφου από την ίντα, όπως αναφέρθηκε η κυρία Σαϊφή από το ΕΛΚ, έχει κάνει μια ε, ε, σύνταξε ένα κείμενο. Ε, εγώ θα, λάβω, θα βάλω μείον σε ορισμένες ε, παραγράφους. Δεν είναι ότι είμαι εντελώς κατά. Αντιθέτως, θεωρώ ότι ορισμένες από αυτές τις παραγράφους είναι τόσο πλούσιες και πολλές φορές επαναλαμβάνονται κάποια σε σχέση με αυτά που έχω στην έκθεση μου. Επίσης, το αριθμό 16 προτείνω μια χωριστή ψηφοφορία. Όχι γιατί είμαι κατά των μικροπιστώσεων, διότι καλύπτονται απλώ αυτά τα θέματα ε, στο κείμενό μου, το βασικό. Επίσης, εφιστώ την προσοχή για χωριστή ψηφοφορία που ζήτησα στην παράγραφο 20, την αρχική μου. Και έχουμε τροπολογία 119. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε από όλου του ιδιώτε και το χώρο της βιομηχανία να αναλάβουν την ευθύνη τους όσον αφορά κάποιες βασικές αρχές αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τους Ευρωπαίους αλλά για όλους και αυτό το λόγο σδίδιτσα για αυτή τη λέξη μια χωριστή ψηφορία. Και μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 21 τη δική μου και για την 24 όπου προτείνω όπου η παραγράφος θα είναι ως εξής to urge the EU and other donors not to facilitate or to contribute να απέχει από τη διευκόλυνση τη συμβολή στην ανάθεση εφορη γη σε χώρε και περιοχέ, όπου υφίσταται επιστηστική ανασφάλεια για άλλου σκοπούς εκτός από την παραγωγή τροφίμων και να δημιουργήσει βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση τη γη και των πόρων. Υπάρχουν και κάνα δύο άλλες χωριστέ ψηφοφορίε σε σχέση με προφορικέ τροπολογίε. Ε, αυτά τα έλαβα νωρίς το πρωί. Θα κάνω αυτό τον κατάλογο, θα τον ετοιμάσω και φυσικά ε, περιμένουμε ανυπομονώ μάλιστα για την ψηφοφορία του απόγευμα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμβάλλαν για αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι μαζί από κοινού θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σφένσον. Όντως ήταν μια απόφαση που ελήφθη το πρωί στους συντονιστές οι, πράσινοι το εστίασαν που είναι απόντε στο άλλο. Καλώ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Τώρα έχω την ε, ευχαρίστηση να καλωσορίσω την ε, Επίτροπο για τις κλιματολογικές αλλαγές. Δεν έφτασε ακόμα. Θα δώσουμε πέντε λεπτά. Ή όχι. Δεν είναι ακριβώς η ώρα, 11.30. Ε, βέβαια. Απ' τη μια αργούμε, αργήσαμε και απ' την άλλη είμαστε νωρί το πρόγραμμα. Ε, ζητήσαν κάτι πράσινοι, οι πράσινοι δεν είναι εδώ. Θα πρέπει κανεί να ξέρει τι θέλει τέλο πάντων. Όταν ζητάει κανεί ένα θέμα για την ημέρησα διάταξη, τουλάχιστον να είναι παρόν. Τέλο πάντων, α δώσουμε πέντε λεπτά τώρα στην Επίτροπο να έρθει. Ε? Alors, il y a des disputes comme ça en Θα ήθελα να σας πω το εξή. Έγραψε σήμερα το πρωί η γραμματεία ότι οι πράσινοι ζήτησαν ανταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες ε, Σβένσον, αλλά τώρα μου λένε ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι μου λένε. Αλλά αλλάζουν τα πράγματα κάθε δύο λεπτά. Δεν το έπανε, το ζήτησαν οι πράσινοι. Λυπάμαι κύριε Σβένσον, εγώ έτσι ε, είδα ότι το ζήτησαν οι πράσινοι. Οι πράσινοι τώρα λένε ότι δεν το ζήτησαν, τώρα σταματώ γιατί εκνευρίζομαι. Παρακαλώ, ας οργανωθούμε καλύτερα. Εκνευρίστηκα λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και σταματώ. Έχω την ευχαρίστηση να παρουσιάσω, να καλωσορίσω την Επίτροπο Κόνι Έντεγκορντ για τις κλιματολογικές αλλαγές. Ε, δεν το πρόφερα καλά. Έντεγκορντ έπρεπε να πω. Γαλλίδα είμαι και ξέρετε πως είναι οι Γάλλοι με αυτά. Η κυρία Έντεγκορντ δέχτηκε την πρότασή μας να έρθει εδώ να γίνει ανταλλαγή απόψεων οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ένα σημαντικό θέμα. Ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα, καταστροφές, μεγάλες καταστροφές για τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες και το θέμα είναι σημαντικό, έχει μεγάλη έκταση. αυτό το θέμα στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες δεν περιορίζεται εκεί όμως, είναι και σφαιρικό και θα χρειάζεται δική μας συμμετοχή και άλλοι να συμβάλλουν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, διότι έχουμε να κάνουμε με το κοινό καλό της ανθρωπότητας και για μας τους ίδιους. Κάποια μέρη στον κόσμο πλήττονται ιδιαίτερα με αυτές τις αλλαγές και είναι πιθανόν ότι οι αλλαγές που γίνονται θα αρχίζουν να εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και φυσικά με επιπτώσεις όσον αφορά την μετανάστευση πληθυσμών οι κλιματικές αλλαγές ε, δε, επεκτείνονται, εντείνονται και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο η, η αρχή όσον αφορά το να συμβάλλει κανείς χρηματικά είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται σε διεθνές επίπεδο και δι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο μας και κυρίως η Επιτροπή μας πρέπει να κάνει τα μέγιστα. Κυρία Επίτροπε, ε, να μην εκπλήσεστε, διότι είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, ε, αρχές ενάντια σε οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί και έχουμε, δίνουμε έμφαση όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης και ξέρω ότι αυτό είναι και δική σας επιθυμία. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε φυσικά ότι, ότι οι, οι χώρε χώρες ζητούν και βοήθεια να τις υποστηρίξουμε διότι ε, υπάρχουν μαζικές επιπτώσεις όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Κύριε Επίτροπε, εσείς και εμείς από κοινού πρέπει να προχωρήσουμε στην ίδια κατεύθυνση και να κοιτάξουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια ε, και μια πορεία από κοινού. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα αμέσως το λόγο στην κυρία Head Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μου δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις ε, για την ε, κλιματική αλλαγή όσον αφορά την ανάπτυξη. Όπως ακριβώς είπε η Πρόεδρος, η κλιματική αλλαγή και η εξάλληψη της φτώχειας είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει από κοινού. 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας ε, και δεν καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αισθητέ ε, και ήδη επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και όλο και περισσότερο, όπως είπε η Πρόεδρος, θα βλέπουμε επιπτώσεις και σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Ήδη σήμερα οι κλιματικές αλλαγές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων μεγάλος αριθμός και μεγάλη ένταση φυσικών καταστροφών, έλλειψη νερού και τροφίμων. Αυτά είναι απλώς λίγα παραδείγματα. Το κατόφλι της αύξησης ε, θερμοκρασίας των δύο βαθμών φαίνεται ότι θα το φτάσουμε αν δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Πέραν από το κατόφλι αυτό υπάρχει ένας πολύ ψηλότερος κίνδυνος ε, να συμβούν αμετάκλητες καταστροφές που θα οξύνουν ε, τα προβλήματα έλλειψης φαγητού και νερού, αυξάνοντας περισσότερο τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει διασύνδεση αυτών των θεμάτων και όταν το συζητάμε με εκπροσώπους των αναπτυσσομένων χωρών, όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό αυτό το θέμα. Ενώ πριν από 5-10 χρόνια δεν το αναγνώριζαν αυτό το θέμα. Τώρα έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν και πολλοί υπουργοί και κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες τώρα πια βλέπουν ότι υπάρχει ανάγκη να μπουν και τα θέματα κλιματικής αλλαγής στην αναπτυξιακή τους πολιτική και στρατηγική. Όπως γνωρίζετε, το φθινόπωρο θα γίνει μία εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και τη δουλειά που θα ακολουθήσει μετά το 2015. Παράλληλα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, πάλι υπάρχει αυτή η προθεσμία του 2015. Το, στο Παρίσι το 2015 θα θέλαμε να κλείσει συμφωνία για το κλίμα. Δηλαδή το 2015 είναι ένα έτος ορόσημο, γιατί παράλληλα δύο πολύ σημαντικά θέματα προχωρούν και πρέπει να φτάσουν στο να δώσουν καρπούς και πέρυσι τον Ιούνιο η διάσκεψη του Ρίο 20 τόνισε την ανάγκη να υλοποιήσουμε δράσεις ε, σε μια πράσινη οικονομία. Αυτό το οποίο ήταν περιβαλλοντική συζήτηση στη μία πλευρά και αναπτυξιακή συζήτηση στην άλλη πλευρά, όλο και περισσότερο γίνονται δύο συζητήσεις που διασυνδέονται. Λίγες μέρες ε, μετά το συμβιβασμό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είπε και η Πρόεδρος, γίνεται αυτή η συζήτηση και ε, σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για το κλίμα. Μας ενδιαφέρουν παράλληλα και άλλοι τομείς όπου βρίσκονται σε διασύνδεση το κλίμα και η ανάπτυξη. Κατανοώ τις ανησυχίες σας ε, που εκφράστηκαν και προς την επιστολή σας, τη διακομιτική επιστολή προς ε, τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία αποδεκτή προς όλα τα θεσμικά όργανα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι από τις διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα βγει κανείς απόλυτα ικανοποιημένος. Η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί μια αύξηση περίπου 3% του τίτλου ε, του κεφαλαίου ε, για ε, την ανάπτυξη σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό και υπάρχουν νέες δραστηριότητες για το Ταμείο Ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί στον προπολογισμό όλων των κρατών μελών, άρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξήσουν το δικό τους αναπτυξιακό προϋπολογισμό για να μπορέσει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της και όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια γενικά και όσον αφορά τη χρηματοδότηση για θέματα κλίματος αφετέρου. Το 2020 μάλλον στην Κοπενχάγη όλοι οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι δεσμεύονται ε, για τον προϋπολογισμό 100 ε, εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τη χρηματοδότηση του κλίματος και πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, θα τηρήσουμε αυτό το στόχο. Θα πρέπει να εξετάσουμε και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Ξέρω ότι η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, προγραμματίζει κάποια έσοδα από το μελλοντικό φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να τα χρησιμοποιήσει για αναπτυξιακούς σκοπούς. Επίσης, θα έχουμε ε, τέλη που θα δημιουργηθούν από την αρχή ορυπαίνων πληρώνει στον τομέα της ναυτιλίας και αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για το κλίμα. Ακόμη πρέπει να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιδιωτικές πηγές ε, για, την, ε, για τις κλιματικές δράσεις. 100 δισεκατομμύρια ε, ετησίως για όλο τον πλανήτη δεν είναι κάτι που μπορεί να βγει από τον δημόσιο προϋπολογισμό, πρέπει να βρούμε πιο καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης. Αναγνωρίζω ότι η μείωση της φτώχειας ως βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κάτι το αναμφισβήτητο. Και δεν ήρθα εδώ για να σας πω τι ποσοστό θα έπρεπε να δοθεί από το Αναπτυξιακό Ταμείο ή από το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας ε, για το κλίμα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές προτεραιότητες ε, για την ε, υγεία, για την παιδεία κλπ. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια και η στρατηγική για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής για το κλίμα δεν είναι χωριστά. Είναι αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοενισχυόμενα εφόσον δράσουμε έξυπνα. Επομένως, δεν θα πρέπει η χρηματοδότηση του κλίματος να ανταγωνίζεται άλλους αναπτυξιακούς στόχους. Πρέπει όμως εντελώς ειλικρινά να πούμε ότι ένα αίτημα όπως η έκθεση Μπέρμαν πέρυσι τον Ιούνιο να είναι ε, πάνω από το 0,7% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, πόσο πιθανό είναι να γίνει δεν θα συνυπολογίζουμε την χρηματοδότηση για το κλίμα μέχρι να φτάσουν όλα τα κράτη-μέλη στο 0,7% ή θα ήταν πιο δίκαιο να πούμε ότι θα είναι πρόσθετο στην επίσημη νοτιξιακή βοήθεια που δίδεται σήμερα. Οπότε θα πρέπει να συνυπολογίζεται και να γίνεται αποδεκτό ως κάτι το πρόσθετο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό πίσω από την έκθεση Μπέρμαν, αλλά αν δείτε αυτά που προγραμματίζουν τα κράτη-μέλη, Βλέπετε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει φτάσει το στόχο του 0,7% εδώ και χρόνια, αλλά γνωρίζουμε το να φτάσουμε στο 0,7% για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πολλές προκλήσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση ε, για τους στόχους μας, για το κλίμα, για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί πριν από τέσσερα χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πρόσθετο θα πρέπει να σημαίνει πρόσθετο σε σχέση με αυτά τα οποία πληρώνουμε τώρα, όχι πρόσθετο σε σχέση με το 0,7% επίσημης αναπτυξιακή βοήθειας, παρότι όπως είπα καταλαβαίνω το σκεπτικό. Τέλος, θέλω να πω ότι έχω ακούσει και τις χώρες εταίρους μας ε, που εξελίσσουν ε, το σκεπτικό τους γιατί όπως σας είπα βλέπουν τις συνθήκες από την κλιματική αλλαγή και καταλαβαίνουν την ανάγκη να έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική συνεπή με τη στρατηγική μας για το κλίμα. Στην Τόχα το Δεκέμβριο άκουσα εκπροσώπους ε, από την Αφρική, από την Ασία, από τη Λατινική Αμερική να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια για να αυξηθεί η αντοχή των πληθυσμών τους, να προστατευτούν οι πληθυσμοί που ζουν κοντά σε επικίνδυνες ακτογραμμές, να τους βοηθήσουμε με τεχνικές ε, που ε, δημιουργούν λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και ο Υπουργός Ανάπτυξης του Μπαγκλαντές, παραδείγματος χάρη, είπε ότι η προσαρμογή για το κλίμα έχει άμεση σχέση με την επιβίωση της χώρας του και ζήτησε τους ηγέτες παγκοσμίω να λάβουν άμεσα δράση ούτως ώστε να μειωθούν και οι μεταναστευτικές κινήσεις και η ανάγκη μετατόπισης πληθυσμών. Ο Πρωθυπουργός της Ζουαζιλάνδης ε, στην Τόχα μίλησε εκ μέρους όλων των ηγετών της Αφρικής όταν είπε ότι θέλει να δίνεται συγκεκριμένη βοήθεια για δράσεις προσαρμογής και τεχνολογίας και είπε ότι και αυτό συνδέεται με το συμφέρον της χώρας του και των χωρών εκ, των, εκ μέρους των οποίων μιλούσε και ο Υπουργό Περιβάλλοντος της Τζαμάικα είπε ότι η χώρα, η χώρα του χάνει 2% του ΑΕΠ ετησίως λόγω τυφώνων, πλημμυρών, ε, ξηρασίας και αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί, όπως είπε, για να βελτιώσουν την παιδεία μας, την υγεία μας και τις υποδομές μας. Ξέρω ότι σήμερα ε, ή μάλλον συζητήσατε την έκθεση του ΦΑΟ για τη Γεωργία. Αυτή η έκθεση λέει ότι η πρόσφατη επισητιστική κρίση και οι αλλαγές του κλίματος έχουν θέσει τη γεωργία ως προτεραιότητα της διεθνούς ημερήσιας διάταξης. Βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται η σύγκληση των στόχων, δηλαδή εξάλληψη της φτώχειας και αηφόρος γεωργία ε, και ε, όπως λέει η έκθεση του ΦΑΟ η εξάλληψη της φτώχειας θα βοηθήσει τις επενδύσεις στη γεωργία και θα βελτιώσει την ποιότητα των επενδύσεων. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε όταν μιλάμε ε, για δράσεις για το κλίμα που θα πρέπει να ενταχθούν σε όλες τις πολιτικές και να γίνουν ε, έξυπνες ως προς το κλίμα οι επενδύσεις στη γεωργία. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, τη δημιουργία αποβλήτων, να αποφύγουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έξυπνες τεχνικές. Και όταν μιλάμε για υφόρο ανάπτυξη, αυτό εννοούμε. Όταν επενδύουμε να γίνεται αυτό με έξυπνο τρόπο, ώστε να κάνουμε κάτι καλό και για την τοπική οικονομία και παράλληλα και για την παιδεία παρέχοντας ενέργεια, κάνοντας όμως κάτι το οποίο δεν ε, θα ε, είναι αντίθετο με αυτά που κάνουμε σε σχέση με τους στόχους μας για το κλίμα. και το Μπαγκλαντές έχει ε, κάποιες ε, πολιτικές για το κλίμα και ο Μπαρόζο που είχε πάει σε νήσους του Ειρηνικού πριν από ένα χρόνο είχε πει ότι θέλουμε οι επενδύσεις μας να γίνονται με πιο έξυπνο τρόπο ε, και οι άνθρωποι επιτόπου θέλουν οι επενδύσεις μας να έχουν μεγαλύτερη απόδοση γιατί θα γίνονται με πιο έξυπνο τρόπο. Μέσα λοιπόν στην αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να ενταχθούν οι στόχοι για το κλίμα. Δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. μα ενδιαφέρουν και τα δύο εκ παραλλήλου γιατί είναι αλληλοσυνδεόμενοι στόχοι. Με κάθε ευρώ που δαπανούμε θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αμέσως θα δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Μίτσελ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε για την παρουσίασή σας και για τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Η πρώτη είναι η εξής. Σωστά νομίζω λέτε ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το 0,7%. Αν πρέπει όμως βασιζόμενοι στο παρόν επίπεδο των δαπανών πιστεύετε ότι θα μπορούμε ε, θα είναι ε, σωστό να βάλουμε εδώ, να υπολογίσουμε τα ποσά που χρειάζεται να βοήθεια ή θα πρέπει να τα θεωρήσουμε χωριστά. Ένα άλλο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος είναι το εξή. Έχουμε έναν ειδικό ε, πρόσωπο στη Γενέβη, στο πλαίσιο του ΙΕ, για την μείωση κινδύνου. Και ε, για την υποστήριξη της αντοχής, της ανθεκτικότητας σε κάποια θέματα είναι παρεμφερείς θέσεις που έχετε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή οι... κάποιοι κίνδυνοι δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά εν μέρη. Αυτό όμω το οποίο στα... στον ονομάζεται DRO, και αυτό το οποίο κάνει ο ειδικό επίτροπο και αυτό που κάνετε εσεί για την ε, χρησιμοποίηση αυτής της τριπλής προσέγγισης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πώς μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Κύριος Γκέρενς. Να, να υπογραμμίσω τον θυσιασμό με τον οποίο η κυρία Πέτροπος παρουσίασε τις απόψεις της. Ε, ε αλλά παρόλα αυτά εγώ να πω ότι δεν συμφωνώ και τόσο πολύ διότι είμαι σε στην αντιπολίτευση τα λέγαμε σε σχέση με αυτά που είπε. Με όλο το σεβασμό. Καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα ε, γίνεται για τον αγώνα αυτόν που αγωνίζεται για τις κλιματολογικές αλλαγές. Εγώ θέλω να δούμε την ουσία και τη βοήθεια που δίνει η Επιτροπή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπατε, δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει κανείς με δημόσιους, δημόσια κονδύλια όσον αφορά την ανάπτυξη. Η συνένεση που έχουμε στην Ευρώπη αναφέρει την δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη. απο, αποκλειστικά από δημόσια κονδύλια δηλαδή γίνεται βοήθεια. Εσείς λέτε ότι είσαστε μια χώρα η οποία ξεπέρασε ήδη και το 0,7% το δέχομαι και εγώ είμαι από μια χώρα η οποία ε, έχει ξεπεράσει αυτό το ποσοστό, το 0,7. Δεν μιλάμε για τις χώρες οι οποίες πετύχαν ήδη το στόχο. Τι γίνεται με τις άλλες χώρες. Εκτός από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, φυσικά, που δεν μπορούν να κάνουν την ίδια προσπάθεια. Αλλά ε, κάτω από το 0,7% είμαστε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ε, άρα τελειώνουμε με αυτό το στόχο. Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει μια σαφίστατη διάκριση ανάμεσα ε, στα, μέσα που έχουμε για την ανάπτυξη και τα συμπληρωματικά μέτρα. Ότι ξεπερνάει το θέμα ε, που έχει να κάνει με τον αγώνα κατά των κλιματολογικών ε, αλλαγών θα είναι κάτι, θα είναι κάτι συμπληρωματικό. Αν τώρα υποχωρήσουμε τώρα πραγματικά τι κάνουμε, τα παρατάμε. Υποχωρούμε σε ένα στόχο στο οποίο υπήρξε μια συνένεση το 2005 για την ανάπτυξη. Και επανειλημμένα έχει θυχθεί αυτό το θέμα και εδώ και αλλού στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ένα πράγμα το οποίο αναφέρεται εδώ και καιρό και συνεχώς. Λοιπόν, αν κάνουμε αυτό που λέτε, τι κάνουμε, δημιουργούμε μια ρήξη. Ε, εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος πάνω σε αυτό. Δέχομαι ότι, ότι είπατε πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Μα ζητούν να χρησιμοποιήσουμε ένα 100 του ΑΕΠ για να μπορέσουμε προλάβουμε φέρει μια μεγάλη καταστροφή και σε αυτό το 1% αυτό πρέπει να γίνει μέσα από δημόσια κονδύλια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ε, εδώ πέρα και η ευθύνη που έχουν να κάνουν και οι ιδιωτικοί πόροι. Υπάρχει το joint implementation που λέμε. Είναι μέτρα ε, που έχουν να κάνουν από αυτούς οι οποίοι έχουν ε, προκαλέσει, ε, έχουν μολύνει, έχουν ρηπαίνει. Υπάρχουμε δηλαδή την αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Έχουμε το στόχο του 0,7% και τις ανάγκες που απαριθμίσατε και, και ήταν σωστό αυτό που κάνατε να τις απαριθμίσετε ανάμεσα στη διαφορά, η μόνη διαφορά ανάμεσα σας και εμάς λέω τώρα λέω εμάς γιατί υποθέτω ότι η Επιτροπή μας εδώ ε, παραμένει σαφή στους στόχους της η, δηλαδή η μόνη μας διαφορά είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να βρούμε δηλαδή και αλλού κάποια μέσα είπατε ότι θα πρέπει να πετύχουμε το 0,7% πριν να χρηματοδοτήσουμε. Όχι, μην λέμε ότι έχουμε ένα μέρος στο οποίο χρηματοδοτούμε για την αγώνα κατά της χρηματολογικής αλλαγής και απ' την άλλη έχουμε την δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη που είναι για τον αγώνα κατά της φτώχειας. Είναι δυο τομείς χρηματοδότησης οι οποίοι είναι παράλληλοι. Δεν μπορούμε να τα ε, συμπτύξουμε αυτά και να υπάρχει μια σάφια για το τι ακριβώς ισχύει. Όλα αυτά θα ενταχθούν στα πλαίσια της δημόσιας, των δημόσιων διαπάνων για την ανάπτυξη. Δηλαδή και τον αγώνα για την κατά της φτώχειας και τις κλιματολογικές αλλαγές. Έχουμε και τα κριτήρια της ε, Επιτροπής για την Ανάπτυξη του ΟΣΑ. Η ξέρω ότι ήταν λίγο ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα ποτέ δεν απάντησε με σαφήνεια για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσον αφορά αυτά τα ερωτήματα. Ξέρω ότι αυτό βολεύει τις χώρες μέλη, τα οποία προφτιμούν να είναι σε μια έτσι ε, ομιχλώδη κατάσταση. Γι' αυτό εμείς είμαστε απαιτητικοί. Ίσως να είμαστε ε, αφελείς, ίσως να είμαστε υπερβολικοί, αλλά υποστηρίζουμε αυτή τη θέση διότι ε, ε είμαστε από αυτούς οι οποίοι ε, κάνουμε αυτόν τον αγώνα πάνω στον οποίο υπήρξε μια συνένεση εδώ και 8 χρόνια. Θεωρώ ότι προδίδουμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση πάνω σε αυτό το θέμα. Το τελευταίο στάδιο ε, έχει να κάνει στο λεγόμενο package deal στα πλαίσια χρηματοδότησης 14-2020 ε, όπου ενσωματώνει κανείς τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη γίνεται μια μείωση τις, ε, στις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν, ότι δεν έχει δαπανηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει από τις χώρες μέλη. Και τι βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραδοθεί, το βλέπουμε στο τελευταίο συμβούλιο και βλέπουμε και τις χώρες μέλη να μην συμφωνούν όσον αφορά τους στόχους χρηματοδότηση. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα θεμελιώδε πρόβλημα. Δεν είσαστε υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δει, να καταλήξει κάπου, να, να εκφραστεί κάποιο εξ ονόματι της Επιτροπής, διότι τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ε, διαφορετικά. Θα πρέπει, και χαίρομαι και σας ευχαριστώ που είσαστε παρούσα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Έχω πραγματικά πρόβλημα με αυτό. Δεν υπάρχει, δεν έχει μπει τάξη σε όλα αυτά. Πρόεδρος, πριν να απαντήσει η Επιτροπή και ο κύριος Ντέβα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ γιατί με πάθος υπερασπιστήκατε τη θέση σας και το σέβομαι αυτό. Χρειαζόμαστε, νομίζω, σαφήνεια για τα θέματα αυτά, όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς γιατί ε, υπάρχει κάποια σύγχυση για το πώς εξετάζουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την αλλαγή του κλίματος. Όλο και περισσότερο αρχίζω να νομίζω ότι ο κύριος Γκέρενς και εγώ είμαστε σε ένα συνασπισμό. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει. Όπως οι συνάδελφοι στη Βουλή των Κοινοτήτων συμφωνούν με τους φιλελευθέρους. Εν πάση περιπτώσει. Στην, αλλαγή, στην κλιματική αλλαγή υπάρχουν τρία πράγματα. Πρώτον, Υπάρχει αυτό το οποίο κάνει ο ήλιος. Επί χιλιάδες χρόνια περάσαμε από εποχές των παγετώνων, από θερμές περιόδους, από ψυχρές περιόδους, πράγματα που δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπους. Έχουν σχέση μόνο με εκείνη τη μεγάλη φωτεινή μπάλα στον ουρανό που δημιουργεί και ηλιακές κοιλίδες. Δεύτερον, υπάρχει το επιχείρημα ότι εμείς επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία με αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, οι άνθρωποι. Αυξάνουμε το διοξίδιο του άνθρακος. Και τρίτον, υπάρχει η ρήπανση που έχει οξύτατες επιπτώσεις σε ορισμένα θέματα, τα οποία πολύ συχνά δεν αναφέρουμε καθόλου. Παραδείγματος χάρη, στα Ιμαλάια ε, έχει επιταχυνθεί το λιώσιμο των πάγων ε, τετραπλάσιο, σε τετραπλάσιο βαθμό σε σχέση με οπουδήποτε αλλού λόγω του διοξιδίου του άνθρακος και υπάρχει ε, ένα μια τεράστια πιθανότητα πλημμύρας γιατί οι παγετώνες λιώνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμένετο. Πράγμα το οποίο θα σημάνει και ε, ε, πλημμύρες και ξηρασία και πείνα για ε, τεράστιες ομάδες πληθυσμού. Αυτό δεν συζητήθηκε πουθενά. Ούτε στο Ρίο, ούτε στην Κοπενχάγη, ούτε πουθενά. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι μπορεί να πεινάσουν λόγω αυτού. Σκεφτόμαστε τώρα το πώς θα τιμωρήσουμε τις ε, χρηματοοικονομικές μας υπηρεσίες, διότι οι ρηπαντές ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Γιατί θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο Λονδίνο να φυγεί, επειδή κάπου αλλού κάποιος άλλος μεταφέρει ρηπαίνοντα προϊόντα. μιλάμε νομίζω με τρόπο που δημιουργεί σύγχυση. Το City του Λονδίνου που ελπίζω ότι θα εξαιρεθεί από το φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καλύτερα να εξαιρεθεί διαφορετικά δεν θα μείνει η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει το City να φύγει γιατί κάποιος στην Κίνα έχει σταθμούς παραγωγής ενέργειας με κάρβουνο που ε, δημιουργεί συνθήκες ρήπανσης σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν κάπως θα πρέπει να τα συζητήσουμε από κοινού, διαφορετικά δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα αφήσω την Επίτροπο να απαντήσει και μετά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων με βάση στον πειρασμό να μπω σε μια μεγαλύτερη συζήτηση για τη στρατηγική του κλίματος γενικότερα, αλλά θα προσπαθήσω να εστιαστώ στο βασικό θέμα της συζήτησής μας σήμερα. Να πω όμως ε, προς τον αξιότιμο κύριο Βουλευτή ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν συζητάμε τον άνθρακα που ρηπαίνει τα Ιμαλάια. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε σε πολλές πρωτοβουλίες για τις διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε συνεργάζεται και προσπαθούμε να κάνουμε έρευνα αντί να περιμένουμε να γίνει κάτι από μόνο του. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την εθάλη, το μαύρο άνθρακα. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσω προς τον κύριο Μίτσελ. Η Επίτροπος Γεωργίευα και εγώ και το τι κάνουμε στη Γενέβη όπως είπατε. Η Επίτροπος Γεωργίευα και εγώ προσπαθούμε η κάθε μία από την πλευρά της να το προσεγγίσει και συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ε, το σκεπτικό του πολιετούς πλαισίου χρηματοδότησης όσον αφορά το κλίμα ε, δείχνει ότι θέλουμε να μην απομονώσουμε τη στρατηγική για το κλίμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε σε μια γωνίτσα χωρίς κανένα συντονισμό. Μπορεί να το ακούσατε και από την ίδια την Κρυσταλίνα Γεωργίευα όποτε επισκέπτεται χώρε μετά από φυσικές καταστροφές είτε στο μάλι είτε στην αϊτή όπου και αν πηγαίνει έρχεται και μου λέει κάθε φορά μέσα σε αυτές τις φυσικές καταστροφές πάντοτε κάπου υπάρχει κάτι σχετικό με το κλίμα και όταν θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ανασυγκρότηση βλέπουμε ότι πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή κάπως πρέπει να βρεθεί τρόπος να μπει μέσα στον προϋπολογισμό σε όλα τα σημεία. Πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά και για τις μεταφορές και για τη γεωργία και για την ενέργεια. Για όλα τα θέματα πρέπει να έχουμε κατά νου την κλιματική αλλαγή. Και έχουμε συμφωνήσει τώρα με το Συμβούλιο ότι 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ιχνηλάσιμος. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε εκ των υστέρων ότι όντως έχει ληφθεί υπόψη το κλίμα σε οποιαδήποτε μέτρο λαμβάνεται. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και με τον συνάδελφο Πίμπαλξ έχουμε καλή συνεργασία και ένας από τους τομείς προτεραιότητας για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και για τον ίδιο τον κύριο Πίμπαλξ είναι η Αφρική και η ενέργεια για την Αφρική πάλι στο ίδιο σκεπτικό δηλαδή ότι για να εξαλειφθεί η φτώχεια πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην ενέργεια και γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο πιο φιλικό προς το κλίμα και περισσότερο για φόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε μαζί και να μην ξεχωρίζουμε καν κάθε χαρτοφυλάκιο. Και το γραφείο στη Γενέβη αυτό κάνει, ρωτάει ο κύριος Μίτσελ. Κάνουμε συναντήσεις, απαντάει η Επίτροπος. Δεν λέω ότι κάνουμε καθημερινές συναντήσεις, αλλά έχουμε συναντήσεις και αυτοί έχουν επιχειρήματα όσον αφορά την ε, αντοχή για το κλίμα και είχαν ε, εκδώσει την έκθεσή τους με τη συνδυασμένη γνώση που υπάρχει για αυτό το θέμα. Και η Κρυσταλίνα Γεωργίευα ήταν παρούσα και εγώ προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε σε όλους αυτούς τους τομείς γνώσης. Προς τον κύριο Γκέρενς για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Προσωπικά εγώ υπερασπίστηκα πάρα πολύ στεναρά το 0,7% και μέσα στην Επιτροπή ε, τονίζω ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε γίνει τόσο φτωχοί που να μην μπορούμε ε, να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε λάβει δέσμευση ότι θα κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επομένως, αυτό το οποίο λέω δεν είναι ότι δεν μας νοιάζει το 0,7% και στη διακήρυξη του Ρίο υπήρχε ότι η Ευρώπη έχει και διατηρεί και επαναδιακηρύσει τη δέσμευσή της για το 0,7% επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και της χρηματοδότησης για το κλίμα. Όταν ε, βλέπουμε την πραγματικότητα ότι η Ευρώπη δεν είναι στο 0,7% και από τα στοιχεία που έχω από τον προϋπολογισμό των κρατών μελών ε, βλέπω ότι ακόμη και οι χώρες που ήταν πολύ περήφανες γιατί παρήχαν το 0,7% τώρα παρουσιάζουν κάποια μείωση. Βλέποντα λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάσταση, εδώ έχουμε δύο γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Από τη μία πλευρά πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε συζητήσεις σε εσωτερικό επίπεδο και να συζητάμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε το 0,7% επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Η άλλη γραμμή είναι το τι θα λένε οι εκτός Ευρώπης όταν λένε ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση για το κλίμα να είναι κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό το οποίο ήδη είχατε τις δεσμεύσεις του 2009. Εκείνοι λένε ότι αυτοί που βρίσκονται από την άλλη πλευρά, δηλαδή αυτοί που, είναι, που είναι, λαμβάνονται στη βοήθεια, θα μετρήσουν το αν η Ευρώπη κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό που έκανε το 2009. Δηλαδή θα πρέπει να δίνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που τότε δίναμε. Δίκαιο είναι και αυτό. Ε, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα γιατί μας λένε οι απ' ότι πρέπει να δώσετε το 0,7 και μετά θα δούμε ε, τι δίνεται για τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Μπορούμε τότε να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη όντως δίνει αυτά που έχει υποσχεθεί για το κλίμα. Για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνολικά ισχύει το ότι το κλίμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσουμε σε μια γωνίτσα και αφού τελειώσουμε με την πολιτική για τη γεωργία, αφού τελειώσουμε και με την πολιτική για τις μεταφορές θα πει κάποιος «Α, και το κλίμα, και αυτό πρέπει κάπου να το βάλουμε». Πιστεύω ότι πρέπει την πολιτική για το κλίμα να την εντάξουμε σε όλες τις άλλες πολιτικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην πολιτική κάθε κράτους μέλους ε, χωριστά πρέπει το σκεπτικό για το κλίμα κατά τον ίδιο τρόπο να ενταχθεί και στις αναπτυξιακές μας στρατηγικές. Και εδώ δεν μιλάμε για το μέγεθος του προϋπολογισμού. Αυτό είναι απλώς ένας έξυπνος τρόπος να κάνουμε αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι είπατε κύριε Γκέρενς ότι αν η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ήταν μόνο εξάλληψη της φτώχειας και εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε γιατί εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη και η παιδεία τι είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για τα 27 κράτη-μέλη. Πολλές δραστηριότητες και θα σας έλεγα ότι αν πάτε σε ένα χωριό στην Τανζανία με ένα έργο ε, όπου έχουμε βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στις καλύβες τους και αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για το τοπικό σχολείο και για τους δασκάλους και για τους μαθητές και για τις γυναίκες και για τα κορίτσια και ούτω καθεξής. Για μένα αυτό είναι καλή αναπτυξιακή πολιτική γιατί έχει εντάξει και την οπτική γωνία του κλίματος. Θα ήταν ανόητο να μην κάνουμε τέτοιου είδους προγράμματα με τρόπο που θα προάγει και τη στρατηγική για το κλίμα, παράλληλα δηλαδή με την αναπτυξιακή μας βοήθεια. Είναι σημαντικό και το 0,7, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε μια κατάτμιση των πολιτικών μας. Αντίθετα θα πρέπει να τη συντονίζουμε. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η Αιθιοπία. Αν δείτε την αναπτυξιακή στρατηγική της Αιθιοπίας και τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της φτώχειας, η ενέργεια και η προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και όλο και περισσότερο προς τα εκεί θα κινούμεθα, γιατί πιστεύω ότι οι έξυπνες αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενσωματώσει και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Και τέλο, σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, πιστεύω, ελπίζω ότι τώρα θα μπορέσουμε να σταματήσουμε να συζητάμε τους καινοτόμους χρηματοδοτικούς πόρους. Η ναυτιλία, οι αεροπορικές μεταφορές, κάποια μόνιμα έσοδα θα πρέπει να ε, κατευθύνονται και προς την ε, στρατηγική για το κλίμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και να το βάλουμε στα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και νομίζω ότι πρέπει πιο συγκεκριμένα να το αναφέρουμε το 2015 στο Παρίσι. Να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχόμεθα. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Κόρτες Λάστρα κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα και σεβόμενος την άποψή σας. Όπως κατανοείτε, η βιομηχανική πολιτική, η ΚΑΠ, η πολιτική έρευνας, καινοτομίας, ενεργειακή επασχόληση στην ευρωπαϊκή κοινότητα, πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν μια νέα πολιτική. Μιλούμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Και θα προσθέσω και το εξής. Η πολιτική κλιματικής αλλαγής η διεθνούς συνεργασίας που μέχρι τώρα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συμβολική για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για το δικό σας το θέμα, την κλιματική αλλαγή. Όταν λέτε ότι σε κάποια μέρη στην Αφρική ε, κάνετε κάτι με τα φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά ούτε καλύτερες πολιτικές. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να κάνουμε μεγάλα πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν έχουμε ε, την άποψη ότι όλα θα πρέπει να προέρχονται για όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές από τα ίδια κονδύλια και από την ίδια χρηματοδότηση. Είδατε ότι πριν από μερικέ μέρε μειώθηκε ο κοινοτικό προπολογισμό. Είδατε ότι κάποιε χώρε όπω η δική μου ε, περιέκοψε κονδύλια για θέματα συνεργασία. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν το υποστηρίζω και ποτέ δεν το υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια μέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να περάσουμε από τον, το, το, το ίδιο σημείο. Αυτό, το περίφημο 0,7%. Αυτό είναι κάτι με το οποίο, εάν θέλετε, δεν συμφωνούμε. Και βεβαίως συμφωνούμε με την τόσο μεγάλη περικοπή η οποία έγινε σε επίπεδο ε, πολιτικής συνεργασίας, σε επίπεδο υπουργών, ε, όπως αποφασίστηκε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω το εξής, ότι Βεβαίω θα πρέπει να συνδυαστούμε, βεβαίω θα πρέπει να συνεργαστούμε και ο κύριο Μίτσελο είπε, και αυτό είναι πρωτοαρχική σημασία, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του μέλλοντο και για να έχουμε μια κοινή πολιτική. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι στην επιτροπή δική μα ένα από του στόχου είναι στα πλαίσια του 7% διαφωνεί απόλυτα με αυτό το οποίο ε, έγινε με τις περικοπές. Και θα πρέπει και εσείς να εκφράσετε την ε, πλήρη αντίθεσή σας για τα περικοπή των κονδυλίων, για την ε, πολιτική της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι το θέμα σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Εδώ και 10 μέρες, ο στόχος του 0,7% επιβεβαιώθηκε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που έγινε για το επόμενο πολιετές για το προϋπολογισμό 2014-2020 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Γκάρενς. Ε, δεν ξέρω τι αξίζει αυτό που είπατε. Η πρακτική ό, μας δείχνει το αντίθετο. Ε, δηλαδή διατρανώνουν κάτι αλλά κάνουν το αντίθετο. Τέλος πάντων. Ε, θα πρέπει να μην υποχωρήσουμε και να μην προδώσουμε τους στόχους μας. Ξέρω η κυρία ότι έχει ένα αληθινό πρόβλημα. Όλα όσα έχει πει για τις ανάγκε χρηματοδότηση είναι ακριβέστατα. Έχουμε μια συζήτηση και έχουμε μια διαφορά όταν μιλάμε για στόχους και μέσα. Εγώ συμφωνώ με τους στόχους. Δεν συμφωνώ μαζί σα όσον αφορά τα μέσα και τα μέσα χρηματοδότηση συγκεκριμένα. Μια διευκρίνηση επίσης Όσον αφορά τις πολιτικές, συμφωνώ με τη δική σας προσέγγιση. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός με τις πολιτικές που δεν μας οδηγεί πουθενά. Δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μου. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι το εξή. Μιλάμε για την ευθύνη που έχουν οι εταίροι στη διαδικασία. Η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει σαν πρώτο στόχο την απάλληψη της ε, φτώχεια, επενδύνοντας σε διάφορε τομεί. Συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να γίνει επενδύση στην ενέργεια. Το ίδιο και για την εκπαίδευση. Συμφωνώ επίση που λένε ότι ε, να δούμε τα θέματα τη διακυβέρνησης και σε θέματα πολιτισμού φυσικά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν για να συμβάλλουμε ούτως ώστε να μειώσουμε τη φτώχεια. Τώρα, εκεί που δεν συμφωνώ, είναι όταν πρέπει να επενδύσουμε κονδύλια, καταρχήν, που έχουν προβλεφθεί για την απάλληψη της στόγιας. Για να γίνονται κάποιες, ας πούμε, ε, σαν αποζημίωση για, λάθη που έχουμε κάνει εμείς. Ε, στην Κοπεχάγη αναφέρθηκε για να γίνει μια πιο ήπια ε, εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, για τις αλλαγές του, τις κλιματολογικές. Τι γίνεται, δηλαδή τι, διορθώνουμε λάθη που έχουμε εμείς κάνει. Αυτά πριν να πάρουμε αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα κονδύλια. Να γίνεται μια σωστή διάκριση. Η ρήπανση έχει να κάνει με την ευθύνη αυτών που έχουν ρηπαίνει και μετά έχουμε το δημόσιο ε, το, το δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάνω σε αυτό και θέλω να συμβάλλω στο να το λύσουμε. Να κάνουμε καταρχήν μια διάκριση λοιπόν ανάμεσα ε, λίγο έτσι να ε, μειώσουμε το θέμα που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις και το θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια αυτό το θέμα για την έργεια είναι συμβατό με την, ε, τους στόχους της ανάπτυξης. Από τη δική μας οπτική γωνία θα πρέπει να δούμε το θέμα στη διάρκεια, μακροπρόθεσμα, όσον αφορά τις πολιτικές για τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν όλα αυτά, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε Le 0,7% on l'a Euh, έχουμε να κάνουμε όμως για τη μείωση του αποτελέσματος, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Εμείς, να σας πω το εξής, είμαστε κατά της ε, χρησιμοποίησης κονδυλίων, δημοσίων κονδυλίων, για τον αγώνα κατά της, των κλιματολικών αλλαγών, όσο δεν έχουμε επιτύχει το στόχο του 0,7%. Παράλληλα, από τη μια πρέπει να γίνει ε, ε, χρηματοδότηση χρήση των δημόσιων κονδύλων και ο στόχος να επιτευχθεί το 0,7%. Υπάρχουν πολλέ χώρε οι οποίε θέλουν να πάνε προ τα πίσω. Κάνουν πίσω. Δεν γίνεται αποδεκτό αυτό. Ακόμα και αν είναι κυβερνήσει που είναι του ίδιου τη πολιτική οικογένεια που ανήκω. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Και οδηγούν και άλλε χώρε σε αυτό. Λένε πολλά για του Βρετανού, αλλά πρέπει κανεί να του υποστηρίξει κανεί σε αυτό το στόχο, στο 0,7%. όχι να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους, τα δημόσια κονδύλια. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους Βρετανούς μόνους πάνω σε αυτό το. Δεν είναι αυτοί που ευθύνονται λοιπόν στην Ήπειρο, εδώ στην, Ευρωπαϊκή Ήπειρο πρέπει να δούμε αυτούς τους υπεύθυνου. Λοιπόν, να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις επενδύσεις για το μέλλον όσον αφορά την ανάπτυξη, για τις αναπτυσσόμενες χώρες για το μέλλον αλλά θα πρέπει όλοι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Το Clean Development Mechanism, Φερρυπίν, είναι ένα μέσον όπου αυτοί που προκαλούν ρήπανση αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν είναι δημόσιοι πόροι. Οι υπεύθυνοι χρηματοδοτούν λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το ενισχύσουμε και αυτό θα μας επέτρεπε να συγκλίνουν οι απόψεις μας. Μη φύγετε ότι θα σας αφήνουμε ε, μόνοι. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και ο στόχος δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί λόγω του ότι δεν έχουν κάποιον ικανότητα να πετύχουν στόχους. Και θα πρέπει πραγματικά όλοι να ανταποκριθούν στους στόχους για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί. Υπάρχουν όλοι οι εταίροι οι οποίοι έχουν υπογράψει και αυτοί θα πρέπει να το δηλώσουν. Η Επιτροπή να είναι ε, σύσσωμη, να εκφραστεί ε, σύσσωμη πάνω σε αυτό και να μην αλλάζουν τα πράγματα όταν μιλάμε με τον Α ή Β Επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ τον κύριο Γκέρονσον. Η κυρία Χέντεγκορ τώρα πάλι το λόγο για να κλείσει. Πρέπει να πω ότι στην Επιτροπή. Πολλοί έχουμε κοινή άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε και τι χρειάζεται να κάνουμε. Και νομίζω ότι εσείς και εγώ μπορούμε να κάνουμε τώρα συζήτηση για το 0,7 και όταν θα πρέπει η κλιματική αλλαγή να επηρεάσει. Δεν είναι θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας αυτό ακούστηκε στο παρελθόν και λέτε και εσείς ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Συμφωνώ, συμφωνώ με το μηχανισμό της ε, καθαρής ανάπτυξης, της ανάπτυξης χωρίς ρήπανση. Κάποιοι από εμά νομίζω ότι προσπαθούμε για αυτά τα θέματα να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο διεθνώς για ασχολούμαι με θέματα συνεργασία σε θέματα τεχνολογιών. Θέλουμε να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές. Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά χρειάζεται ένα διεθνές πλαίσιο για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και διεθνώς με το θέμα κλιματικής αλλαγής. Και η Ευρώπη στην τελευταία σχετική συνάντηση παραδέχθηκε ότι δεν είμαστε ε, σοβαρή, διότι είχαμε και κάποια προγράμματα τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα και θα πρέπει να δώσουμε κάποιες αντισταθμίσεις. Αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε κάπως υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουμε το όρο θέμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία κλειδιά τα οποία θα συζητούν στην επόμενη σχετική διάσκεψη στην κλιματική αλλαγή στη Βαρσοβία παρά το γεγονός ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το τι θα θέλαμε να έχουμε μακροπρόθεσμα, δηλαδή τουλάχιστον 0,7% από την Ευρώπη και από όλες τις χώρες, και στα πλαίσια της χρηματοδότησης, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι με αυτά που κάνουμε ότι τουλάχιστον το δικό μας το κομμάτι ευθύνη, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής το αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σωστά. Στο Μπαγκλαντές είδα ένα από τα καλύτερα ε, προγράμματα παραδείγματος στα πλαίσια της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Δηλαδή σε κάποιες τρομερές πλημμύρες που έγιναν πριν από χρόνια, τι συνέβη. Συνέβη το ότι δεν μπόρεσε κανένα από τα σπίτια να αντισταθεί στο μεγάλο ε, οστικό κύμα της πλημμύρα. Και έτσι είπαμε ότι στην επόμενη φορά ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, πρόνοια ώστε όλοι να ειδοποιούνται με SMS σε περίπτωση πλημμύρας και να πηγαίνουν σε υψηλότερα κτίρια. Αυτά, ώστε να μην έχουμε θανάτους σε τέτοιες Αυτά είναι θέματα συνεργασίες για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις πιο ανθεκτική την αντιμετώπιση. Μαλή τώρα. Βλέπετε τι σημαίνει. Υπάρχουν εξαιτία της αφαιρήμωσης κάποια προβλήματα με τα κοπάδια των αγροτών, των κτηνοτρόφων που πρέπει να πάνε από το βορρά στο νότο, αυτοί του νότου ε, έχουν πρόβλημα διότι άλλα ζώα έρχονται να βοσκήσουν στα δικά τους λιβάδια για τα δικά των δικών τους ζώων. Υπάρχει πρόβλημα την ε, κοτονού και μπορείτε να δείτε ότι πολλές φορές όταν προσπαθείτε να βοηθήσετε ώστε να αναπτυχθεί μία περιοχή θα πρέπει να δείτε και πολλά άλλα θέματα, κυρίως πώς θα επηρεάσουν την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες τα θέματα αυτά της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θέλω εγώ να πω. Περί αυτού πρόκειται. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε από κοινού και συντονισμένα. Δεν είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε ε, κάτι το αρνητικό ή να επιβάλλουμε κυρώσεις σε αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν από τα κράτη-μέλη να επιτύχουν το στόχο αυτό του 0,7% ή να φτάσουν σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Κύριε Γκέρεν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σύντομα, μία πρόταση έχω να σας κάνω και μία ερώτηση να κάνω και ένα σχόλιο. Η πρόταση που έχω να σας κάνω είναι η εξή. Στα πλαίσια του Κιώτο είχαν προβλεφθεί δύο μηχανισμοί ε, διόρθωση. Το μηχανισμό Clean Development και η Joint Implementation, υποκοινού εφαρμογή. Ο μηχανισμός ε, Clean Development αφορούσε τα αναπτυσσόμενες χώρες και έτσι οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούσαν να δαπανίσουν ε, κάποια κονδύλια, βοηθούν οι χώρες και να ξεπεράσει το επίπεδο ρήπανσης. Θα μπορούσαμε μία χώρα του προσαρτήματος 1 στα πλαίσια της joint implementation να τη βοηθήσουμε να εξάγει την τεχνογνωσία και την τεχνολογία της σε μια χώρα επίσης του προσαρτήματος α, ανεπτυγμένη δηλαδή. Είπαμε ότι μπορεί κανείς να μειώσει το χρέος του σε σχέση με το κιότο είναι μόνο όταν αναλάβει να ε, αμβλύνει την ζημία που είχε ε, δημιουργήσει και προκαλέσει εξαιτία της εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρωπο. Αυτά στα πλαίσια της joint implementation, δηλαδή μεταφορά από ανεπτυγμένη σε ανεπτυγμένη χώρα. Τώρα, στα πλαίσια των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει η Κομισιό, γιατί να μην ε, ε, εξουσιοδοτήσουμε τη μεταφορά τεχνολογίας από μία χώρα ανεπτυγμένη προς μία αναπτυσσόμενη. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνει και τον ιδιωτικό τομέα να απομισεί τις ευθύνε του και θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση της κατάστασης και θα επέτρεπε επιπροσθέτως να ε, ενεργήσουμε με ηλεκτρίνεια. Δηλαδή, κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ε, κάποιες βιομηχανίες που ρηπαίνουν αλλά είναι στο ε, προσάρτημα 1 και δεσμεύονται από το πρωτόκολλο του Κιώτο, τις ε, ε, μεταφέρουμε κάπου αλλού και ρηπαίνουν κάποιον άλλο. Έτσι λοιπόν ε, κάνουμε τον ιδιωτικό τομέα της κάθε χώρας μας να είναι πιο υπεύθυνο. Επίσης, είπατε ότι μακροπρόθεσμα ο στόχος για όλους είναι 0,7. Συγγνώμη, δεν είχαμε ε, δεσμευτεί μακροπρόθεσμα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα το 2015. Και εδώ έχετε να κάνετε με άτομα τα οποία είναι έτοιμα για συμβαστική λύση για να μην ε, προδώσουμε, αν θέλετε, αυτό το στόχο. Ο στόχος αυτός του 0,7% επαναλαμβάνω είναι βραχυπρόθεσμος και βεβαίως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι διότι δεν υλοποιείται ο στόχος. Να έρθουν οι ένοχοι. Αυτοί που αναλάβουν ε, δεσμεύσεις και μετά δεν μπορούν να τις υιοθετήσουν. αυτή είναι η υπεύθυνοι. Και δεν το αποδεχόμαστε αυτό. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια αξιοπιστία. και εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι. Να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι. Μπορώ να κάνω το α και μετά να αλλάζω δρόμο. Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την κοινή εφαρμογή του Joint Implementation, είναι κάτι που συζητήθηκε στην Τόχα, γιατί ο ευέλικτο μηχανισμό υπάρχει μόνο για αυτού που δέχτηκαν και μια δεύτερη περίοδο δεσμεύση. Τέλο δεν θα μπω στι λεπτομέρειε τώρα, αλλά η κοινή εφαρμογή του Joint Implementation και για τη Ρωσία και για τι χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση είχε δοθεί, ενώ δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το CDM όμως θα μπορούσε να είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Προσπαθούμε να το εξυγχρονίσουμε, ούτως ώστε να μην, είναι, να μην έχουμε πολλά μεμονωμένα προγράμματα που συνήθως είναι μικρής κλίμακας. Να έχουμε μία μορφή προγράμματος, δηλαδή να πάρουμε ένα ολόκληρο τομέα, μια ολόκληρη χώρα και να τον εξυγχρονίσουμε και να βάλουμε και μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον ε, ε, Clean Development Mechanism, το CDM. Δεν μπορούν από φέτος ε, τον Ιανουάριο να έχουμε τέτοια προγράμματα σε μικρές χώρες αναπτυσσόμενες. Είναι μία από τις προκλήσεις ε, αυτού του μέσου, αυτού του μηχανισμού, ότι το 90% όλων των ε, προγραμμάτων πήγαν σε κάποιες μεγάλες ε, αναπτυγμένες χώρες και προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε και χρειάστηκε και πολλή δουλειά για να μπορέσει να αλλάξει ο μηχανισμός CDM για να κάνει καλύτερα το έργο του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σα υπενθυμίζω ότι εμεί τις τρει συνεχίζουμε με την Επιτροπή ανάπτυξη με την ψηφοφορία και μην ξεχάσετε την κάρτα σα για την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και στο επανειδήν.